στην Αγία Πετρούπολη, όπου εκεί θα προχωρήσουν περαιτέρω οι συζητήσεις όσον αφορά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν 7 ε, ε, προτάσεις ψηφισμάτων που θα ψηφιστούν μετά τη συζήτηση. Και τώρα γυρίζουμε στο επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη που είναι η Βενεζουέλα και ειδικότερα η υπόθεση της Μαρία Λούρντες Αφιούνη. Ο πρώτος μας ομιλητής θα είναι ο κύριος Σάσα Αξέγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με τον ε, Βολβιανό νόμο, ε, έχει φυλακιστεί ε, κύριος, η κυρία Αφιούνη και ο κύριος Τσάβε ζήτησε να της αποδοθεί η μέγιστη τιμή και επίσης να αποφασιστεί μια επιδείνωση μια επιβάρηση της, ε, της ε, ποινής Όλοι έχουν ε, ανησυχήσει με αυτή την υπόθεση. Δεν είναι μονομένη αυτή η περίπτωση κυρίε και κύριοι. Του αντίον δείχνει την αυταρχική στάση μιας κυβέρνησης η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να συλλαμβάνει τους ε, αντιπάλους τους, να κλείνει εφημερίδες, ραδιοφωνικού σταθμούς και ούτω καθεξής, παραβιάζοντας συνεχώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να απελευθερωθεί άμεσα η δικαστής Αφιούνη. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει Κύριε Βέμπερ, για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και πάλι συζητάμε στο Κοινοβούλιο την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Όχι γιατί θέλουμε, αλλά διότι πρέπει. Διότι η κατάσταση δεν βελτιώθηκε από, από το προηγούμενο ψήφισμά μας. Αντιθέτως, η ιδέα του κράτους δικαίου δεν υπάρχει πλέον διότι υπάρχει τόση πίεση στους δικαστές και στο δικαστικό σώμα και υπάρχει παραβίαση πολλών δικαιωμάτων του ανθρώπου από το δικαίωμα ελευθερίας λόγου μέχρι ιδιοκτησίας. Ε, θα πρέπει οι δικαστικές αρχές να είναι ανεξάρτητες όπως και οι δικαστές αλλά ο πρόεδρος Ούγκο Τσάβος απλώς υπαγορεύει μέσω ομιλιών δημοσίων εις τους δικαστές τι θα πρέπει να αποφασίσουν. Και πολλοί δικαστές ήταν θύματα αυτής της διαδικασίας. Ορισμένοι απεμακρύνθηκαν από τις θέσεις τους ή εγκατέλειψαν τη χώρα και η κυρία Φιούνη είναι το πιο κραγγαλαίο πρόσφατο παράδειγμα για την απόφαση την οποία πήρε. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστής να ε, κρίνει την περίπτωσή της αμερόληπτα όταν ε, ε, ο πρόεδρος της χώρας την αποκαλεί κακοποιό και ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να της επιβάλλει τη μέγιστη ποινή. Η Μαρία είναι εδώ και έξι μήνες σε ένα χώρο όπου κινδυνεύει και η σωματική της ακεραιότητα και έχουν ε, κατηγορηθεί για πολύ σοβαρά εγκλήματα. Προσπαθούν λοιπόν να την τρομάξουν και να την εκφοβήσουν και παρακαλώ τον πρόεδρο ε, Τσάβες ε, να ελευθερωθεί. Η κυρία Αλφιούνη θα πρέπει να απελευθερωθεί, αποφυλακιστεί άμεσα και να δικαστεί σύμφωνα με τον νόμο για να μπορέσει να υπερασπίσει τον εαυτό του. Αυτό ε, δεν είναι μόνο σωστό, ορθό, αλλά είναι και μια κίνηση ανθρωπιστικής φύσης. Ευχαριστώ κυρία Ντεκάιζερ, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Στην υπόθεση Μαρία Λούδε Σαφιού στη Βενεζουέλα πρόκειται για καταπολέμηση της διαφθοράς όπως ε, λέει η καταδίκη της ή μια, πρόκειται για μια πολιτική δίωξη σύμφωνα με τους ε, Times. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα. Η ομάδα μου απέσυρε την υπογραφή της ε, από το κοινό ψήφισμα και θα καταθέσουμε ένα δικό μας. Νομίζω ότι υπερφορτώσατε το σκάφος αγαπητή συνάδελφοι και θα ήθελα μέσω αυτής της περίπτωσης την οποία θεωρώ πως θα πρέπει να διευκρινίσουμε και να, δια... και να ρίξουμε άπλετο φως, να καταδικάσουμε όλο το καθεστώς ε, της Βενεζουέλας. Περί τίνος πρόκειται. Η δικαστή Αφιούνη μέσω μιας έκτακτης διαδικασίας αποφυλάκησε έναν τραπεζίτη ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε 27 εκατομμύρια και συνελήφθη. Ε, και Πράγματι, όντως, οι συνθήκες κράτησης είναι φρικτές, είναι απαράδεκτες, όπως και σε όλε τι ε, φυλακέ τη Βενεζουέλα. Αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε εδώ με το θέμα ε, των, σοφρονιστικών καταστημάτων. Θα ήθελα να, να πω το εξή. να υπάρξει μια δίκαιη δίκη με όλες τις εγγύσεις. τη συνέχιση της καταπολέμησης της διαφοράς που υπάρχει στον δικαστικό κλάδο και τον διαχωρισμό του πολιτικού, της πολιτικής εξουσίας από τη δικαστική εξουσία. Όλα αυτά σας τα παραχωρώ, αλλά όλα τα υπόλοιπα σας τα αρνούν. Ευχαριστώ κύριο Ρωμέα Βαϊρουέντα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύμφωνα με τα όσα είπε η κυρία θα ήθελα να πω και εγώ ότι πριν από μερικέ μέρε ζητήσαμε το κατεπήγον και τότε δήλωσα ότι η ιδιαίτερη περίπτωση τη κυρία Αφιούνη άξιζε ιδιαίτερη προσοχή. σω θα έπρεπε να υπάρξει ένα κατεπήγον ψήφισμα μια επιστολή, στην οποία θα μπορούσαν να υποσυμπουράσουν πάρα πολλοί βουλευτέ, ε, κάνοντα έτσι ε, γνωστή την αντίθεσή μας ή και ότι επιθυμούμε να προωθήσουμε αυτή την επιστολή προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας για να επιληθεί το πρόβλημα της κυρίας Αφιούνη. Και αυτό ήταν, αυτή είναι η πρόθεσή μας. Γι' αυτό και εμείς καταθέτουμε ένα ψήφισμα όπου θίξαμε κάποια σημεία τα οποία συμπίπτουν με αυτά τα οποία ακούστηκαν στην αίθουσα. Θα πρέπει λοιπόν να θυμίσουμε το εξή. Ε, αυτό το οποίο είδαμε στην όλη διαδικασία είναι ότι πάνω, εκτό από ένα ψήφισμα σε ένα ζήτημα που αφορά ανθρώπινα δικαιώματα και την ειδική κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζει η δικαστή αυτή τη στιγμή, υπήρξε και ένα ζήτημα που αφορά στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας. Το γεγονός είναι ότι θα έχουμε ε, σε μερικές εβδομάδες εκλογές. Και αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολιτικές επιπτώσεις. Δηλαδή ένα τέτοιο ψήφισμα. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ εδώ στο αν συμπαθώ ή αντιπαθώ τον κύριο Τσάβες. Όχι. Αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί το κοινοβούλιο μας για να κάνουμε προεκλογική εκστρατεία υπέρ της αντιπολίτευσης ε, της Βενεζουέλας. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε ή διαφωνούμε με μια πολιτική, αλλά χρειάζεται πολιτική συζήτηση. Και αυτή δεν είναι μια πολιτική συζήτηση αυτή που έχουμε σήμερα. Θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά να υποθούν σε ένα άλλο πλαίσιο, αλλά όχι τώρα, εδώ. Τα κατεπήγοντα ψηφίσματα έχουν μια συγκεκριμένη, ε, ένα συγκεκριμένο λόγο ύπαρξη και είχατε χρόνο στη διάθεσή για να ε, προβείτε σε αυτές τις ε, καταδίκες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το σκεφτεί το σώμα στο σύνολό του και αυτό προς όφελος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, όλη η δημαγωγία του Προέδρου Οέγκο Τσάβο τη Βενεζουέλα φαίνεται ότι δεν γνωρίζει όρια και τώρα έχει σαν στόχο την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου. Σαν νέο εμπόδιο το θεωρεί για να κατακτήσει την απόλυτη εξουσία. Συλλήψει και τη Μαρία Ζωμιμόρα είναι πολύ ε, η πιο τολμηρή του προσπάθεια να προσπαθήσει να φημώσει τη διαφωνία και να ε, ζητήσει το διαχωρισμό ε, των εξουσιών και να επικρατήσει το Ο ίδιο την, την έχει κατηγορεί ότι έχει δολοκηθεί και είπε ότι πρέπει να φυλακιστεί για 30 χρόνια. Και είπε ότι ο Σιμών Μπολιβόρ θα την είχε εκτελέσει και το καθεστώ του γίνεται όλο πιο δικτατορικό και παρακινεί τη βία με αυτά που λέει. Αν ο Τσάβε συνεχίσει αυτή την συμπεριφορά ε, ατιμωρητή και επειδή είναι δημοφιλής γιατί κατηγορεί τις ΗΠΑ τον υποστηρίζουν πολύ αριστεροί στην Ευρώπη και εδώ ε, αυτό θα είναι κάτι που θα υπονομεύει τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ενώσεως που προσπαθεί να δείξει ότι η Βενεζουέλα οδεύει με ταχύς ρυθμούς προς τον ολοκληρωτισμό. Ευχαριστώ. Είδα μπλε κάρτα από τον κύριο Πόσελτ που φαντάζομαι ότι θέλει να απευθύνει ερώτηση προς τον κύριο Ρωμέβα. Κύριε Ρωμέβα, δεχόσαστε το ερώτημα. Κύριε Σπόσελτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο Ρωμέβα αν ξέρει ότι στην ημερήσια διάταξη δεν υπάρχουν ε, ε, μόνο το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και η περίπτωση Τσάβες είναι περίπτωση δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Κύριε Πόσελ, πρόκειται για θέμα προτεραιοτήτων. Πριν από μερικού μήνε συζητήσαμε το ζήτημα αυτό τη Βενεζουέλα για, σε ένα κατεπήγον ψήφισμα. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρε ποιε είναι οι προτεραιότητε και εάν ε, κρίνεται ότι πρέπει να υπάρχει συζήτηση για την Βενεζουέλα, εντάξει, αλλά αυτό το θέμα δεν έχει καμία σχέση με το ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ πρόκειται για μια στήριξη τη επόλυτευση. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα με του ομιλητέ. Ο κ. Χίγκεν για δύο λεπτά μικρόφωνο ο κύριος Χίγκινς. Okay. Okay. Uh, Αυτό το ψήφισμα που υποτίθεται αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα εκθέτει μια τεράστια υποκρισία ανάμεσα στα δεξιά κόμματα του Κοινοβουλίου. Διότι πραγματικό στόχος δεν είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά να προωθηθεί η πτώση της κυβερνήσεως του Γκοτσάβες της Βενεζουέλα να δοθεί βάση για τα δεξιά κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα και που ελέγχει όμως μεγάλο τμήμα των μέσων ενημέρωσης που είναι ιδιοκτησίας ιδιωτικής και βιομηχανίας και γές και υποστηρίζει εκείνου που προσπάθησαν να κάνουν πραξικόπημα πριν από 10 χρόνια. Η κυβέρνηση Τσάβε έλαβε διάφορα προοδευτικά μέτρα που βελτίωσαν τη ζωή των πλέον φτωχών τμήματων τη κοινωνία και του λαού. Αυτό σημαίνει ότι ο Τσάβε ήταν εναντίον των νεοφιλελευθέρων πολιτικών που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ ΕΕ προσπαθούν να επιβάλλουν σε πολλέ χώρε τη Λατινική Αμερική πολιτικέ όπω η απελευθέρωση, η απορρίθμιση, η ιδιωτικοποίηση, ε, των οικονομιών τους που πρωταρχικά ωφελούν τις μεγάλες υπερεθνικές εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή την εκστρατεία που προσπαθεί να δείξει σαν τέρα στον Τζάβες. Εγώ θα έλεγα ότι η Τζότζια Φιούμι και όλοι οι φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αξιοπρεπώ και θα πρέπει η δίκη του να είναι δίκαιοι. Έχω στις φίλου μου στο σοσιαλισμό ρεβολουσιονάριου συναδέλφου σοσιαλιστέ στη Βενεζουέλα που έχουν σοβαρά προβλήματα με κάποιε πτυχέ των πολιτικών του Τσάβε. Αυξάνονται οι τάσει για γραφειοκρατία και σταλινιστική τάση κατάχρηση και της αριστεράς και του εργατικού κινήματο. Θέλουμε περισσότεροι πόροι του ιδιωτικού τομέα στη Βενεζουέλα να μπουν στο δημοκρατικό έλεγχο και διαχείριση των εργαζομένων που θα είναι βάση για τη δημιουργία ε, θα δημιουργηθούν υπηρεσίε που θα αλλάξουν τη ζωή τη πλειοψηφία του λαού τη Βενεζουέλα και θα σταματήσουν τα φρικτά προβλήματα όπω είναι η φτώχεια και η εγκληματικότητα, αλλά θα παρέχονται και η πλήρη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλου. Ευχαριστώ τους, ο κύριος Σόνιξ, τους μεμονωμένους ομιλητές, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε αυτή την αίθουσα ε, ε, μας τίθε το ερώτημα όπως και στις εκλογικές περιφέρειές μας πόσο αποτελεσματική είναι η δραστηριότητά μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι έχουμε κομμουνιστές συναδέλφους οι οποίοι θεωρούν ότι μπορεί κανείς να ρίξει μια κυβέρνηση με, την, ε, με τις δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά θα ήμουν ευτυχής να ισχύσει κάτι τέτοιο δηλαδή τα καθεστώτα αυτά στη Ρωσία ή αλλού να μπορούν να καταργηθούν με δηλώσει απλώ. αλλά πριν από δύο μήνες είχαμε πει τα ίδια δεν ήταν ούτε ο χρόνο ούτε ο χώρος να συζητήσουμε ε, την Βενεζουέλα πρέπει όμως να προασπίσουμε τα, ανθρωπίνα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ασχέτω ε, των ε, συμπαθειών μα. ο πρόεδρος Τσάβες και το κρατικό, ο κρατικός του μηχανισμός ε, ε, είναι αντίθετος του ε, υπερασπιστές της δημοκρατικής αντιπολιτεύσεως και πέραν της κυρίας Αφιούνη θέλω να απευθυνθώ στην είπα το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να κάνει έκκληση στη Βενεζουέλα και να καταγγείλει την έλλειψη νομιμότητος μέρος αυτής της προσπάθειας. Χαίρομαι που ασχολείται με αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα και που υψώνει τη φωνή του κατά των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα. Έτσι δε περαιτέρω θα καλώ την κυβέρνηση Βενεζουέλας να σεβαστεί το λαό της Βενεζουέλας καθώς και τις διεθνείς, το Διεθνή Χάρτα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να υπάρξει πραγματική δημοκρατία στη χώρα και κράτους δικαίου και να γίνονται σεβαστά. Η περίπτωση αυτή που συζητούμε υπενθυμίζει δυστυχώς την αρνητική στάση της Βενεζουέλας έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κράτηση της Αφιούνη είναι παραβίαση των ατομικών της δικαιωμάτων και σοβαρή απειλή για την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα. Ευχαριστώ. Και τώρα η διαδικασία προσέλκυσης προσοχής της Προέδρου, Catch και έχω περισσότερες αιτήσει για παρεμβάσεις από ό,τι θα μπορέσουμε να καλύψουμε τελικά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η κυρία Κόχολα είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, συζητήσαμε και πριν από έξι μήνες για τα προβλήματα δημοκρατίας στη Βενεζουέλα και ιδιαιτέρως για τις κακές εξελίξεις εις ε, την ε, τοποθέτηση της κυβέρνησης ενάντια στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης τα οποία αποκλείονται, αποκλείονται όπως και διάφορες ιστοσελίδες αλλά στον τομέα αυτό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και ο πρόεδρος επισήμως κατηγόρησε την δικαστή να φιώνει και τη χαρακτήρισε ως κακοποιό. Πιστεύω λοιπόν ότι οι δημοκρατικές αρχές πρέπει να τη χάνουν σεβασμού στη χώρα αυτή και η ελευθερία απόψεως και εκφράσεως πρέπει επίσης ε, να προωθηθούν όπως και η δημοκρατική εξέλιξη υπό ελευθέρων εκλογών. Ευχαριστώ. Κυρία Μακοβάη. Ε, <clears throat> η δημοκρατία στη Βενεζουέλα κινδυνεύει και θα ήθελα να προσθέσω και μια άλλη υπόθεση. Η κυβέρνηση περιόρισε την ελευθερία του λόγου και πιέζει και ελέγχει την κοινωνία των πολιτών. Προσπάθησε η Βενεζουέλα το 2010 να τροποποιήσει το σχέδιο ψηφίσματος για τη συμμετοχή τη κοινωνίας των πολιτών στην ε, διοργάνωση των στην οργάνωση των Αμερικανικών κρατών ήθελε να εφαρμόζεται το κρατικό δίκαιο η Βενεζουέλα και αυτό δημιουργεί κακό προηγούμενο κινδυνεύει όλη η περιοχή. Παρόμοια ρήτρα στην ρήτρα εφαρμογή τη αμερικανική ρήτρα τη σύμβαση αυτή χρησιμοποιήθηκε από τη Βενεζουέλα για να μην, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να μην ανακοινώνουν τι παραβιάσει των δικαιωμάτων στη χώρα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν την κοινωνία των πολιτών στη Βενεζουέλα και θα πρέπει να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ τι επικείμενε κοινοβουλευτικέ εκλογέ. Η νομιμότητα ε, του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντική όταν επιδεινώνεται κατά στη δημοκρατία. Και εγώ θα θενώσω τη φωνή μου για την απελευθέρωση τη δικαστού. Ευχαριστώ κυρία Κρετού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρετή. Θα ήθελα να πω για μία ακόμη φορά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντα ήταν προτεραιότητα για μας, οπότε είναι φυσικό να ανησυχούμε για την κατάσταση αυτή που επικρατεί και τις συνθήκες τις οποίες λαμβάνουν χώρα αυτές οι δίκες και το καθεστώς των κρατήσεων. Θα πρέπει τελικά να, είναι, να επικρατήσει μια η δικαιοσύνη στη δίκη αυτή θα γίνει στη Βενεζουέλα σύμφωνα με το κράτος δικαίου και ταυτόχρονα δεν νομίζω ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται τέτοιες περιστάσεις που δεν ξέρουμε τόσο καλά σαν πρόσχημα για να επεμβαίνουμε στην εσωτερική, στα εσωτερικά της χώρας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολάσιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφραστώ. Ε, όντως εκπλήσωμε για τον τρόπο με τον οποίο ο Τσάβες εξασκεί την εξουσία ή στην Βενεζουέλα ε, θυμίζει την Ανατολική Ευρώπη πριν από την πτώση του τείχους η κυρία Φιούνη κρατείται ε, και ε, δεν υπάρχει ελευθερία λήψεως αποφάσεων βλέπετε ότι η δικαστική αρχή δεν είναι είναι ανεξάρτητοι και ο, η Βενεζουέλα και ο Τσάβες ε, καταστρέφουν τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω το λόγο για την ε, Βενεζουέλα και για την παραβίαση των δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Μάλλον δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι και η τελευταία. Θα ήθελα να αναφερθώ. Τι προηγούμενε φορέ αναφερόμουν σε δημοσιογραφικέ πηγέ. Σήμερα αναφερόμουν σε, θα σε κάποιου πολίτε που θέλουν να ζουν ελεύθερα ανθρώπου ε, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν τι δουλειέ του, ε, τι εργασίε του, τι περιουσίε κλπ. Για πολλούς στο παρελθόν η Βενεζουέλα ήταν μια χώρα υποδοχής. Δυστυχώς σήμερα η ελευθερία έκφρασης αλλά και άλλες ελευθερίες και δικαιώματα αποτελούν παρελθόν. Σήμερα μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και παραβίαση αυτών. Θα θέλα να υποστηρίξουμε την ε, δικαστή Αφιούνη και όλους όσοι ε, δρούν υπέρ της ε, ελευθερίας στην Βενεζουέλα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό, σας ευχαριστώ. Εδώ τελειώνει το η διαδικασία κάτσου και θα ζητήσω από την Επίτροπο να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τροπή ιδίω παρακολουθεί εκ του σύναγκης τα τεκτενόμενα στην Βενεζουέλα και Φυσικά συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην αίθουσα αυτή σχετικά με την κράτηση της κυρίας Μαρία Λούρδε αφιούνη. μετά από τις δηλώσεις της ε, βενεζουαρινής κυβέρνησης. Είναι γνωστό ότι η ομάδα των Εθνών σχετικά με τις αυθαίρετες κρατήσεις ε, χαρακτήρισε την κράτηση της κυρίας ε, Αφιούνη ως ε, μια προσπάθεια ε, που πλήττει την δικαστική ανεξαρτησία. Και δημιουργεί ένα κλίμα φόβου στο δικαστικό σώμα αλλά και στους ε, δικηγόρους και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παρακολεί, την απόδοση δικαιοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιτακτική η άμεση αποφυλάκησή της. Η Διαμερικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέδωσε δήλωση υπέρ της ε, κυρία Αφιούνη και ζητάει την προστασία της ομαρική τη ακαιρεότητα αλλά και τη μεταφορά τη σε μια πιο σίγουρη φυλακή. Όπως ακούστηκε εδώ συνεχίζει να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της ε, φυλακής ε, σε μια φυλακή όπου όπου κρατείτε όπου οι συνθήκες κράτησης είναι αυτές οι ψήσεις ασφάλειας Τα θέματα αυτά εξετάστηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου με τις ε, αρχές της Βενεζουέλας και οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι αυτή η κράτηση είναι σύμφωνη με την νομοθεσία της Βενεζουέλας, αλλά θεωρούμε πως αυτές οι δηλώσεις ε, είναι εσφαλμένες και μας προβληματίζουν. Ε, δυστυχώς βλέπουμε ότι έχει προκύψει ε, μια πόλωση πολιτική ε, εκλογές του Σεπτεμβρίου θα επηρεαστούν από αυτές τις ε, συνθήκες και αυτό το οποίο θέλουμε να ζητήσουμε είναι οι εκλογές να διεξαχθούν δίχως οχλής απειλές και εκφοβισμό των, ε, του πληθυσμού και του σεβασμού των ελεύθερης έκφρασης και του κράτους δικαίου. Εμείς επιθυμούμε να βγει ενισχυμένη η δημοκρατία στην Βενεζουέλα μετά από αυτές τις εκλογές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Δεν μπορώ να δεχτώ μπλε κάρτα παρά μόνο για άλλο μέλος. Έχουμε 7 προτάσεις